άρθρο 6 ε, έμαθα ότι δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από την διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών ως προς την Γιούρη για καταεξιοδότηση πράξης. Εάν μέσα σε 24 ώρες δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες, θα εγκρικεί διαδικασία διαφορετικά θα γίνει ψηφοφορία. Υπάρχει η σχετική σύσταση στην ιστοσελίδα μας.